πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και δίκαιος και ισότιμος κατημερισμός των ωφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους στην Ένωση. Το λόγο έχει η κυρία Μπελιέ για τέσσερα λεπτά ως εισηγήτρια για να μας παρουσιάσει το κείμενό της και γνωρίζετε ότι θα έχετε και δύο λεπτά στο τέλος για να κλείσετε. Αν χρησιμοποιήσετε λιγότερο χρόνο τώρα, θα μπορέσετε στη δευτερολογία σας να τον εξαντλήσετε. Έχετε αμέσως το λόγο κυρία Μπελιά, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μετά από 20 χρόνια διεθνών διαπραγματεύσεων, το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Διεθνή κοινότητα έκαναν ένα βήμα για την προστασία της βιοπικιλότητας με προσέγγιση δυναμική και το πρωτόκολλο Ναγκόγια για μια δίκαιη και ισότιμο καταρμερισμό των ωφελών από την χρήση. Θέλουμε να μεταφέρουμε το πρωτόκολλο Ναγκόγια και να επιτρέψουμε στην Ένωση να το επικυρώσει πριν από τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών 2014. Αυτό εντάσσεται μέσα σε μια δυναμική προοπτική των υποχρεώσεων μας. Η βιολογική ποικιλότητα που είναι το φυσικό μας κεφάλαιο. Ο Πρόεδρος. Συγγνώμη, οι συνάδελφοι διερμηνείς με ειδοποιούν ότι τρέχετε υπερβολικά. Παρακαλώ να μιλάτε πιο αργά. Έτσι κι αλλιώς είμαστε αρκετά λίγοι για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το χρόνο και να σας ακούσουμε. Και θα τελειώσετε την παρέμβασή σας. Δεν χρειάζεται να τρέχετε. Ακόμα και αν ξεπεράσετε κατά τη το χρόνο σας. Να αρχίσω λοιπόν πιο ήρεμα. Συνεπώ, η έκθεση που θα ψηφίσουμε αύριο είναι να μεταφέρει το πρωτόκολλο Ναγκόγια και να επικυρωθεί, ώστε να επικυρωθεί πριν από την επόμενη διάσκεψη των ΗΠΑ το 2014. Το σχέδιο κανονισμού είναι μέσα στα πλαίσια τη δυναμική των υποχρεώσεων μα και δεσμεύσεων ω προ την βιολογική ποικιλότητα που είναι το φυσικό μα κεφάλαιο. Η κρίση, η απώλεια των ζώντων οργανισμών επιτρέπει εν τρίτον των ειδών απειλούνται και πολλά οικοσυστήματα υποβαθμίζονται. Έχουμε μια κρίση των ζών των οργανισμών σημαντικότητα και έχει συνέπειες σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές που κάθε μέρα έχουν ε, μεγάλο τίμημα, όλο και μεγαλύτερο. Η έκθεση ενέχει πρωταρχική σημασία στις σχέσεις με τους διεθνείς εταίρους. Το πρωτόκολλο είναι η θέσπιση ενός συστήματος για υφόρο ανάπτυξη για όλους, για το βορρά, τον νότο, ενισχύει ε, τον σεβασμό, τον αμοιβαίο μέσα σε ένα πλαίσιο ε, κρίσης οικονομικής, ηθικής, πολιτικής στην Ευρώπη και διεθνώς. Επίσης έχει ευρωπαϊκή πολιτική σημασία στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την βιοπικιλότητα. Η Ευρώπη επευλήθη ως σημαντικός εταίρος, επέτρεψε σημαντικά βήματα προόδου απαραίτητα για την υιοθέτηση του πρωτοκόλου Ναγκόγια. Από την ψηφοφορία την αυριανή ε, θα εξαρτηθεί η παρουσία της Ευρώπης στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και ο ρόλος και η θέση της Ευρώπης στην διεθνή σκηνή στον τομέα του περιβάλλοντος. Θα εξαρτηθεί επίση επίσης το μέλλον του ευρωπαϊκού οικονομικού μοντέλου, ένα πιο ίσο, πιο ε, δίκαιο ε, μοντέλο αηφόρο. Έχουμε διακυβεύματα βεβαίως στην προστασία της βιοπικιλότητας, αλλά πολλοί τομείς οικονομική και έρευνας, πολλοί πληθυσμοί που εξαρτώνται από την βιοπικιλότητα ε, επηρεάζονται. Θα πρέπει να έχουμε κανόνες σαφείς και δίκαιους για όλους τους Ευρωπαίους χρήστες για να ενθαρρύνουμε την έρευνα, να ενθαρρύνουμε τις εταιρείε μας και να προ προωθήσουμε την καινοτομία σεβόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από το πρωτόκολλο εξαρτάται η εμπιστοσύνη με τους διεθνείς εταίρους και μπορεί να χάσουμε όλη την αξιοπιστία που επί χρόνια οικοδομούμε με συμμαχίες και συνεργασία. Και αυτό όχι μόνο στις διαπραγματεύσεις για τη βιοπικιλότητα, αλλά επίσης και σε άλλες διεθνείς συναντήσεις. Αν είναι απούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση από το πρωτόκολλο του Κιώτο και το κλίμα, τι θα σκεφτούμε. Το ίδιο ισχύει για την βιολογική ποικιλότητα και το πρωτόκολλο Ναγκόγια. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο μας καλούν να προωθήσουμε την διαδικασία για να τηρήσουμε τη διεθνή ατζέντα. Ωστόσο, δεν αρκεί το πρωτόκολλο Ναγκόγια αν δεν έχουμε έναν ευρωπαϊκό κανονισμό που να σέβεται τους στόχους του πρωτοκόλλου. Γι' αυτό εργαστήκαμε όλοι μαζί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τους συναδέλφους και όδης εισηγητές για τη συνεργασία τους. Εργαστήκαμε μαζί για να έχουμε μια θέση στερεά, σοβαρή ε, και ισορροπημένη που βελτιώνει την πρόταση ε, της Επιτροπής και ενισχύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλοί συνάδελφοι υποστήριξαν την έκθεση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αυτό ισχύει για το μηχανισμό νέων χρήσεων, ούτω ώστε να μην υπάρχει κανένας, καμιά ανταγωνιστική ανισορροπία. Να έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο για την βιοπικιλότητα και ζητούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια νομοθεσία δυνατή, ισχυρή, και να θέσει τέρμα στην βιοπειρατεία όπως την ονομάζουμε. Ο καθένας από εμά έχει αναλάβει τις ευθύνες του και σας ζητώ αγαπητοί συνάδελφοι να εγκρίνετε αύριο την έκθεση έτσι όπως υιοθετήθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και να μου επιτρέψετε να αρχίσω την διαδικασία διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο για να επιταχύνουμε την επικύρωση του ε, πρωτοκόλου Ναγκόια. Ευχαριστώ, Σαντρίν. Το λόγο έχει ο Επίτροπο Ποτότσινο για να μα παρουσιάσει τη θέση Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. Ευχαριστώ. Αξιότιμε Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Σαντρίν Μπελιέ για ε, την ευρυθή τη εργασία σε αυτή την πολύ σημαντική πρόταση. Το ίδιο ισχύει και για τους σκιώδεις εισηγητές, καθώς επίσης και τους εισηγητές των επιτροπών που γνωμοδοτούν. Είμαι ευγνώμων που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πολλά από τα μέλη του αφιέρωσαν τόσο πολύ χρόνο στην πρόταση ε, του κανονισμού αυτού. Γνωρίζω ότι στι εσωτερικές σας συζητήσεις για το θέμα αυτό και στα διαδικαστικά ε, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Αυτό δεν με εκπλήσει, διότι το θέμα αυτό πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και του δίκαιου και ισότιμου καταμερισμού των ωφελών ε, είναι δύσκολο θέμα. Από την άλλη, μάλλον το πόλιο αφενός αφορά την βιοπικιλότητα και το σεβασμό των κυρίαρχων δικαιωμάτων άλλων κρατών, αλλά υπάρχουν και τα δικαιώματα των αυτοχθόνων και ηθαγενών κοινοτήτων που έχουν παραδοσιακή γνώση σε σχέση με τους γενετικούς πόρους. Από την άλλη πλευρά όμως έχει επιπτώσεις και για οικονομικές αξίες τις οποίες είναι προσιλωμένοι και έχει μεγάλο συμφέρον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα να είναι το περιβάλλον πρόσφερο για την καινοτομία, να προστατεύονται επιχειρήσεις κτλ. Οι διαπραγματεύσεις του πρωτοκόλου της Ναγόγια χρειάστηκαν πάρα πολύ χρόνο και ε, πραγματικά υπάρχει μια ισορροπία εκεί μεταξύ των διαφόρων ε, ενεχομένων συμφερόντων. Το γνωρίζω αυτό από πρώτο χέρι, διότι ήμουν παρόν, όπως και πολλοί από εσάς. Τώρα βεβαίως έχουν τελειώσει οι διαπραγματεύσεις και θα πρέπει να ε, εφαρμόσουμε τα συμφωνηθέντα. Είμαι πεπισμένος ότι η έκθεση που σας παρουσιάστηκε και στην οποία αύριο θα ψηφίσετε θα αποτελέσει μια γερή βάση για διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων επί του θέματος αυτού. Ακόμα και αν πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάποια σημεία. Η επιτυχία της ε, νομοθετικής αυτής διαδικασίας και εν ώψη των ευρωεκλογών ε, ε, ε, είναι κρίσιμη και θα εξαρτηθεί πολύ από το αν θα δοθεί η εντολή στην κυρία Μπελιέ για να αρχίσει η διαδικασία. Ο χρόνος είναι χρήμα γιατί υπάρχει και προθεσμία τον Ιούλιο για την θέση σε ισχύ του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια και η επικύρωση είναι μια διαδικασία μακροχρόνια και επίπονη δεν επιτρέπεται καμία καθυστέρηση. Ε, κάθε εβδομάδα που περνάει, κάθε μήνα που περνάει μα χρειάζεται για να προχωρήσουμε προ μια συμφωνία μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για να ολοκληρώσουμε και να καταλήξουμε στο κείμενο των διαπραγματεύσεων. Εάν εμεί, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη δεν είναι σε θέση να ε, κυρώσουν εγκαίρω, δεν θα συμμετέχουμε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων στην πρώτη συνάντηση τον Οκτώβριο του 2014. Δεν θα έχει θέση ουσιαστική παρά μόνο παρατηρητή θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί δικαίωμα ψήφου. Αυτό επί της ουσίας θα έχει σοβαρές επιπτώσεις για την επιρροή που μπορούμε να ασκήσουμε εμείς ε, για τις βασικές διατάξεις του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια και πώς θα εφαρμοστούν αυτές. Είναι ε, σοβαρό μειονέκτημα και εις βάρος των κοινοτικών συμφερόντων και μάλιστα ευρωπαϊκών εταιριών αυτή η αδυναμία μας να συμμετέχουμε και είναι και εμπόδιο για τις εταιρείε και τη δραστηριοποίησή τους και πολλές χώρες μπορούν να απαγορεύσουν στους Ευρωπαίους ερευνητές και στη βιομηχανία την πρόσβαση καν στους γενετικούς πόρους. Ορισμένοι πιστεύουν ότι δεν θα υπάρξει καθόλου τέτοια νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν καθυστερήσουν τα πράγματα. Ορισμένα κράτη-μέλη ε, προχωρούν στη δική τους νομοθεσία ενδιάμεση και μεταβατική με αποτέλεσμα τελικά να προκύψει μια κουρελού από κοινοτική νομοθεσία. Αυτό δεν είναι ε, ούτε προς όφελος της εσωτερικής αγοράς, ε, ούτε υπάρχει αρκετή σαφήνεια και ε, προβλεψιμότητα των καταστάσεων. Ξέρετε ότι ήταν πακέτο το πρωτόκολλο της Ναγκόγια. Οι Ευρωπαίοι χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξασφάλιση πρόσβασης σε γενετικούς πόρους σε χώρες αναπτυσσόμενες που είναι πλούσιες σε βιοπικιλότητα και σε γενετικούς πόρους. Θα πρέπει και εμείς λοιπόν να ανταποκριθούμε ε, στις υποχρεώσεις μας να συμμορφωθούν οι χρήστες των γενετικών πόρων σε ευρωπαϊκό έδαφος έτσι ώστε οι χώρες που παρέχουν τους γενετικούς πόρους να έχουν ένα μέρος του ωφέλους, το μερίδιο που τους αναλογεί. Σήμερα συζητούμε ένα κανονισμό που έχει στόχο να δημιουργηθεί αυτό ε, το νομικό πλαίσιο για συμμόρφωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δεν καταφέρουμε να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν οι τρίτες χώρες να αρχίζουν να μας θεωρούν ως ε, μια δικαιοδοσία ανασφαλή ή μη συνεργάσιμη και δεν θα θέλουν να μας ε, δίνουν πρόσβαση στους γενετικούς πόρους σε Ευρωπαίους χρήστες. Ε, έτσι λοιπόν οι κολλησιεργίες και η αναβολή της κύρωσης του πρωτοκόλλου του Ναγκόγια είναι εις βάρος των κοινοτικών συμφερόντων. Επιπλέον, αν δεν έχει κυρωθεί εγκαίρως το πρωτόκολλο θα υπάρχουν πολύ σοβαρές αρνητικές Στι ε, στις διεθνείς υποχρεώσεις μας καθώς επίσης και στο κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και στην αξιοπιστία και στην επιρροή της στην επόμενη ε, σύνοδο των μερών της σύμβασης καθώς και σε άλλα θέματα και φόρα που συνδέονται με ζητήματα περιβάλλοντος. Αξιότιμο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορεί να έχουμε διαφορετικά διαφορετική θεώρηση μάλλον για διάφορα θέματα στα θεσμικά όργανα και δεν είναι σπάνιο. Γι' αυτό υπάρχει ο τριμερής διάλογος για να επιλύονται τα εκκρεμή ζητήματα για να βρίσκεται κοινό έδαφος. Και εγώ είμαι αισιόδοξο ότι μέσω των, των τριμερών διαλόγων θα μπορέσουμε να βρούμε ε, συμβιβασμούς ε, αποδεκτούς με αποτέλεσμα και έκβαση καλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ερευνητές της, τις εταιρείες της και βεβαίως και για τη βιοπικιλότητα. Θυμάμαι ακόμα πάρα πολύ καλά πολλούς από εσάς ε, που με ενθουσιασμό ε, υποστήριζαν ε, θέμα αυτό στην Αγγόια για να προχωρήσουμε στο πρωτόκολλο και στην ενίσχυση της βιοπικιλότητας. Όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, η κοινωνία των πολιτών και οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων συνεργάζονται για αυτό τον ευγενή και αξιόλογο στόχο το 2010. Τώρα έχει έρθει η ώρα να θυμηθούμε ξανά αυτές τις μέρες και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και πάλι για να συμφωνήσουμε εγκαίρως για τον κανονισμό αυτό ε, και είναι χωρίς καμιά αφιβολία προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων ημών καθώς επίσης και της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας που δεν είναι λιγότερο σημαντικό. Θα πρέπει διεθνώς να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης, για ένα λεπτό, η Δόκτωρ Γκρέζ. Καλησπέρα σε όλους. Αγαπητοί συνάδελφοι, στο ίδιο ενέθουσα τα χέρια μας σηκώθηκαν χωρίς αμφιβολία για να πέσει το θέμα της ε, βιοπειρατείας και αυτός ο νέος ε, νέου τύπου υπεριαλισμός ε, ε, να, να, να, πάψει. Όχι στην συγκέντρωση των γενετικών πόρων στα χέρια κάποιων εταιριών των βιομηχανοποιημένων χωρών ε, με τις συνέπειες που γνωρίζουμε. Είπαμε όχι στην εμπορία, όχι στην χρήση γενετικών πόρων που παράνομα έχουν αποκτηθεί. Το πρωτόκολλο της Ναγκόγια είναι σήμερα το μόνο εργαλείο για να καταπολεμήσουμε την βιοπειρατεία. Και το να ε, πολεμήσουμε τη βιοπειρατεία σημαίνει να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών, να διατηρήσουμε την ε, τροφική ασφάλεια. Η Κομισιόν μας άκουσε με το ένα αυτή. Η εξηγήτριά μας έκανε εξαίρετη δουλειά, μας προτείνει ένα ισορροπημένο κείμενο. Να είμαστε λοιπόν συνεπείς με τους εαυτούς μας και αύριο σας καλώ να υπερψηφίσετε αυτό το κείμενο που μας υποβάλλετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω στην αίθουσα τον κύριο Μποβέ που έπρεπε να γνωμοδοτήσει εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και θα ήταν πάρα πολύ σημαντική η συμβολή του. Ας περιμένουμε, μπορεί να έρθει κατά τη διάρκεια της συζήτησης να του δώσουμε το λόγο. Τώρα για ένα λεπτό η κυρία Λέβιν, εξ ονόματος της Επιτροπής Αλίας, παρακαλώ. Σα Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη Σάντριν Μπελιέ και τον συνάδελφο Ιαν Χάτστον το οποίο η έκθεση υιοθετήθηκε με πλήρη πλειοψηφία στην Επιτροπή Αλίας, που είναι σπάνιο πράγμα, και όλες οι τροπολογίες ε, της ηγήτριας υιοθετήθηκαν κατά συνέπεια από την Ουσίας Επιτροπής. Και τέτοιο είδου συμφωνία ανάμεσα στην Επιτροπή Αλίας και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι ακόμα σπανιότερη. Η γνωμοδότηση του κυρίου Χάζτον ασχολείται με δύο σημαντικά θέματα. Καταρχήν αναφέρεται ρητά στην ανάγκη να συμμετέχουν οι τοπικές κοινότητες και να έχουν ε, σε σχέση με την πρόσβαση. Αυτό υπάρχει στο πρωτόκολλο αλλά λείπει από την πρόταση της Κομισιόν και αναγνωρίζει τη δυνατότητα να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της δράσης ε, εκτός των, στα διεθνή ε, ύδατα, πέρα από τα 200 μίλια δηλαδή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι δύο τρίτα των ωκεανών του κόσμου, το μισό δηλαδή της ε, ε, της υδρογείου σφαίρας είναι εκτός εθνικής δικαιοδοσίας. Ευχαριστώ Ιζαβέλα και τώρα πάμε στους ομιλητές που μιλάνε εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων και πρώτα για δύο λεπτά στο όνομα του ΕΛΚ έχει το λόγο η κυρία Γκουτιέρες Κορτίνες. Χριστίνα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που μιλήσατε ε, και εργαστήκατε ε, σε αυτή την προσπάθεια, κυρίως τη Σαντρίν Μπελιά. Αλλά θέλω να ζητήσω την κατανόησή σας και τη περισυλλογή όλων μας για να προχωρήσει αυτό το έγγραφο. Τι είναι αυτό το έγγραφο. Εντάσσεται σε ένα διεθνές σύστημα. Το εξήγησα και στην ομάδα μου ακριβώς για να μας υποστηρίξουν στο έγγραφο. Γιατί. Διότι στην Ευρώπη Έχουμε ένα κορισμό αυτή τη στιγμή νομοθεσίας. Οι επιχειρήσεις, οι εταιρείες και το σύστημα έχουν μπει σε ένα τεράστιο κορσέ, πάρα πολύ στενό. Το κείμενο αυτό είναι ένα διεθνές κείμενο. Και όπως και τόσα άλλα πράγματα θα πρέπει να το δεχτούμε και να μπούμε σε αυτό το διεθνές σύστημα. Και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πολύ ισχυρή και να είμαι σε θέση και η ομάδα μου να το υποστηρίξει. Καταλαβαίνω ότι είναι σωστό το πρωτόκολλο της Ναγόγια. Είναι σωστό να αποζημιώνονται οι χώρες προέλευσης. Είναι σωστό να υπάρχει σωστή εκμετάλλευση. Αλλά είναι ένα κείμενο το οποίο ακόμα δεν έχει οριμάσει. Είναι άγωνο. Θα πρέπει να ε, βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε τη διαδικασία. Γιατί λείπουν εργαλεία και βάσεις. Τι εννοώ. Τα δικαιώματα. Παράδειγμα, έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις, αλλά πού είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Λείπουν πολλά μέσα. Ας πούμε, η επιστήμη είναι πάρα πολύ σπάνιο μια χώρα να έχει εξαντλητικό κατάλογο όλων των γενετικών πόρων και να ξέρουμε σε ποιον ανήκει κάθε προϊόν πραγματικά ουσιαστικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατή και να ε, ε, το ερευνήσει και να το υποστηρίξει αυτό δημιουργούνται πολλές ε, φρούδες ελπίδες σε πολλούς λαούς. Και επίσης θέλω να πω ότι η ομάδα μου θα υποστηρίξει το κείμενο μόνο εάν ε, ε, βγει η αναδρομική ισχύς. Αλλιώς αν καταψηφιστεί θα φταίνε εκείνες οι ομάδες που δεν θέλησαν να υποχωρήσουν. Αυτό το θέμα της ιδιοκτησίας και της αναδρομικής ισχύω είναι κόκκινη γραμμή. Ευχαριστώ πολύ. Από τους σοσιαλιστές το λόγο έχει ο κύριος Παύλ Πότς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, λέμε ότι ε, δεν είναι για βιοπικιλότητα αλλά για την εφαρμογή του πρωτοκόλου Ναγκόγια, της σύμβαση. αλλά βλέπω ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία ε, με τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν υπάρχει εντολή και δεν έχει επικορηθεί, δεν έχει επικυρωθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του Κοινοβουλίου το πρωτόκολλο της ε, Ναγκόγια. Θα έχουμε την διάσκεψη του 2014, δεν θα έχει επικυρωθεί. Υπάρχουν αρκετές χώρες ε, για να επικυρώσουν το πρωτόκολλο χωρίς εμάς. Ε, δεν είμαστε ίσως στο τραπέζι, είμαστε στο μενού. Με και ασχολούμεθα με όλα τα, τις του θέματα θα συζητηθεί χωρίς εμάς η πρόσβαση για το πρωτόκολλο του Ναγκόγια. Θα χάσουμε κάθε αξιοπιστία που οικοδομήσαμε την τελευταία δεκαετία. Βεβαίως ε, θα υποστηρίξω το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, αλλά καλώ όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν την έκθεση ούτως ώστε να δοθεί η εντολή να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Ε, και αν ε, ορισμένοι δεν ψηφίσουν. Μόνο έτσι θα μπορούμε να διαπραγματευτούμε το καλύτερο αποτέλεσμα με το Συμβούλιο και σε αυτή την περίπτωση θα είμαστε μέρος των διαπραγματεύσεων στην επόμενη διάσκεψη του Οκτωβρίου 2014. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων για δύο λεπτά το λόγο έχει ο κύριος Γκερμπράντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε μετά από 18 χρόνια διαπραγματεύσαν τον Οκτώβριο 2010 είδαμε ξαφνικά μια συμφωνία για το πρωτόκολλο του Ναγκόγια και ήμουν εκεί και είδα τον λευκό καπνό. Το αδιέξοδο ανάμεσα σε αυτούς που θέλανε πρόσβαση στις γενετικούς πόρους και αυτούς που ήθελαν ε, να μοιραστούν καλύτερα αυτούς τους γενετικούς πόρους, ξαφνικά αυτή η αντιπαράθεση λύθηκε. Ε, δεν ξέρω αν είμαστε εμείς, ε, εμείς τα μέλη του Κοινοβουλίου, η Κομισιόν, χαιρετήσαμε αυτή το αποτέλεσμα. Ήταν μια νίκη για την βιοπικιλότητα στο μέλλον, στο μέλλον. Και υπήρχε ακόμα το εμπόδιο της επικύρωσης αλλά νομίζω ότι τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από ό,τι είχαν προβλεφθεί, διότι τις τελευταίες μέρες κυρίως πολλές εταιρείες ε, κινητοποιήθηκαν σχετικά με την χρήση των γενετικών πόρων και φαίνονται ότι τώρα, ε, φαίνεται ότι τώρα έχουν δυσκολίες. Υπάρχει νομική αβεβαιότητα και μήπως πολλοί από αυτούς έχουν ε, ιστεροβουλίες, έχουν δεύτερες σκέψεις για το καταμερισμό των ωφελών αλλά ορισμένα πράγματα είναι σημαντικά. Ο στόχος αυτής της πρότασης είναι οι χρήστες να κάνουν έρευνα και ανάπτυξη για τους γενετικούς πόρους. Οι αγρότες λοιπόν και οι έμποροι δεν είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Οι ε, εξαιρέσεις ε, για καλλιέργειας ε, είναι εξασφαλισμένες και αυτοί. Και αυτό με φέρνει στο σημείο κλειδί και για ορισμένες ομάδες είναι ίσως και η κόκκινη γραμμή σχετικά με την έκθεση αυτή. Είναι οι νέες χρήσεις. Μου λέχθηκε ότι χωρίς να περιλάβουμε νέες χρήσεις αυτό το έγγραφο ε, θα ε, είναι ε, κάτι ε, το άχρηστο, διότι 90% ε, των πόρων έχουν εξασφαλιστεί. Τι θα γίνει με το άλλο 10%, γιατί να έχουμε λοιπόν κάτι τέτοιο. Η ερώτησή μου στην Κομισιόν και θα είναι η τελευταία μου φράση κύριε Πρόεδρε είναι είναι αλήθεια ότι χωρίς νέες χρήσεις δημιουργούμε ίσως κάτι το, κάτι το γραφειοκρατικό ή νομίζετε ότι είναι ένα βήμα πρόοδου για καλύτερη πρόσβαση και καλύτερο καταμερισμό ωφελών και ένα μεγάλο βήμα για την βιοπικιλότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έχουμε και άλλους ομιλητές εγγεγραμμένους ε, που μιλούν εξ ονόματός τους. Ο Ντόρφμαν Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παγκοσμίω είναι ηγέτης στην παραγωγή ε, και στην εξαγωγή σπόρων και ε, δεντριλίων και μικρών φυτών και όχι μόνο μεγάλες εταιρείες που ακούμε πάντα αλλά πάρα πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτές οι εταιρείες θα χαρούν πιστεύω να έχουν σαφείς κανόνες για το πώς θα πρέπει να αποκτούν πρόσβαση στους γενετικούς πόρους γιατί έτσι δημιουργείται ασφάλεια δικαίου και διευκολύνεται έτσι ε, και η πρόσβαση σε νέους γενετικούς πόρους Αλλιώς δεν μπορεί κανείς να, παράγει σπόρους και να κάνει τις απαραίτητες καλλιέργειες. Αλλά δεν θα πρέπει να ε, εισαγάγουμε κανόνες που να κάνουν τα πράγματα πιο αυστηρά ε, σε σχέση με άλλες χώρες του κόσμου. Και θα φύγουν εταιρείε από την Ευρώπη αν γίνει κάτι τέτοιο. Στην κύρωση του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια θα πρέπει να προσέξουμε τα εξής σημεία και στην έκθεση που ψηφίζουμε αύριο δεν θα πρέπει να απαιτούμε κανόνες πέρα από το πρωτόκολλο της Ναγκόγια. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, δεν θα πρέπει να έχουμε αναδρομική ισχύ του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια. Τρίτον, δεν χρειαζόμαστε ένα ιδιαίτερο ταμείο για να μπαίνουν χρήματα και μετά να μην ξέρουμε πού πηγαίνουν. Αλλά να ξέρουμε πού προέρχονται από τις εταιρείε. Τέταρτον, δεν θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες ε, που να αμφισβητούν το προνόμιο των παραγωγών και πέντε δεν θα πρέπει να υπάρχει αλυσίδα ευθύνης πέρα από τον πρώτο παραγωγό. Είμαι πεπισμένος ότι αν επιβάλλουμε αυτές τις πέντε αρχές η εφαρμογή του πρωτοκόλου της Ναγκόγια θα είναι προ όφελο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που παράγουν σπόρους και δεντρίλια στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για δύο λεπτά η κυρία Κρίστα Κλάς. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Η Διεθνή Συμφωνία για το Πρωτόκολλο για αγκόγια είναι οι κατευθυντήριες γραμμές και πρέπει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καλή βάση ε, και δεν θα πρέπει να την κάνουμε πιο περίπλοκη ούτε να την βαρύνουμε ε, με άχρηστη γραφειοκρατία. Πρόκειται και για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε σχέση με τρίτες χώρες και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνάδουν με τη βιοπικιλότητα και τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζουν οι γενετικοί πόροι για την παραγωγή τροφίμων και φυτών. Θα πρέπει η γεωργική έρευνα να υποστηρίζεται γιατί μόνο έτσι ε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις ανάγκες ε, παραγωγής τροφίμων για τον πληθυσμό της γης και για τους γενετικούς πόρους. Υπάρχει κάποια αξία και σημασία ε, για την προστασία των ειδών. Αυτά τα έχει συζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα έχει ε, αναγνωρίσει στο πακέτο για το κοινοτικό δίπλωμα τεχνίας Και στις 10 Μαΐου του 2012 επίσης είχαμε αντίστοιχη απόφαση για τις ευρεσιτεχνίες για τις παραγωγές και τις μεθόδους. Γεωργική καινοτομία είναι αυτό που μας ενδιαφέρει και ταυτόχρονα ε, η χρήση των γενετικών πόρων να είναι και προς όφελος ε, των ε, ιδιοκτητών τους. Αλλά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι αγρότες στο μέλλον αυτές τις πηγές Εγώ ποντάρω ε, σε μία πρακτική και ισορρόπη ε, έκβαση αυτής της υπόθεσης και παρακαλώ να δώσουμε στον Επίτροπο τη διαπραγματευτική εντολή για να παραμείνει η Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις και να μην ληφθούν οι αποφάσεις ερήμην της. Ευχαριστώ. Έχουμε και κάτι Ένα μόνο γεγραμμένο συνάδελφο. Σας θυμίζω ότι έχουμε ένα λεπτό στο Κατσδία έκαστος ο κύριος Πάσκα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό το σχέδιο κανονισμού είναι βασικά η μεταγραφή μιας διεθνούς συμφωνίας στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, το πρωτόκολλο Ναγκόγια, που θα μεταγραφεί είναι σημαντικό εργαλείο κατά της βιοπειρατείας και υπέρ της μεγαλύτερης δικαιοσύνης όσον αφορά τους γενετικούς πόρους και τα έσοδα από αυτούς. Συνήθως όλα αυτά γίνονται ε, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αυτόχθονες λαοί. Βέβαια θα πρέπει να γίνουν και προς όφελος των χρηστών. Θα πρέπει να τονίσουμε μια ισορροπία και τη χρήση των πόρων αυτών ε, από όλους. Γι' αυτό θα πρέπει να τονίσουμε καταρχήν το γεγονός ότι με τις ευρεσιτεχνίες πάντοτε θα πρέπει να δηλώνεται η πηγή του γενετικού πόρου και να αποδεικνύουμε πως οι αυτοί οι γενετικοί πόροι συλλέχθηκαν με νόμιμο τρόπο, πράγμα που θα πρέπει να βοηθήσει την χρήση και, τη, και, καταγραφή των γενετικών πόρων, αν όλα αυτά ρυθμιστούν καλύτερα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ε, ανταποκριθούμε στις ιδέες πίσω από αυτό το πρωτόκολλο. Και έτσι ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις των συναδέλφων, λέει ο Πρόεδρος. Και δίνω το λόγο στον, στον ε, Επίτροπο Ποτότσνικ. Σας ευχαριστώ, δεν θα ακρηγορήσω. Βασικά το ερώτημα που ήταν ε, πολύ ευθύ από τον κύριο Γεμπράντη να απαντήσω. Όχι, δεν είναι ένας χάρτινος τίγρης. Η πρόταση για εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλου ε, σημαίνει εφαρμογή του κανονισμού και νέα χρήση και είναι κάτι το οποίο έχουμε πει επανειλημμένως ε, γιατί η, η Κομισιόν δεν συμφωνεί απόλυτα με αυτό όμως πιστεύω πως ε, η έκθεση αυτή μπορεί να είναι μια βάση για διπλωματεύσεις με τις ε, με τα υπόλοιπα, τους υπόλοιπους θεσμούς. Ε, πιστεύω πως οι θέσεις που υπάρχουν είναι πολύ κοντινές και αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια προσπάθεια ώστε πραγματικά να πετύχουμε αυτή την εντολή σύμφωνα με την οποία θα μπορέσουμε να καθίσουμε γύρω από ένα κοινό τραπέζι και να συζητήσουμε πράγμα. Διαφορετικά θα έχει αυτό τεράστιε συνέπειε ε, που είναι δύσκολο και να τι προβλέψουμε καν. Θα τελείωνα λοιπόν ε, λέγοντας ότι Στι αρχέ του περασμένου χρόνου το Ευρωκοινοβούλιο παρότρινε την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για την ε, ε, μεταγραφή του πρωτοκόλου όσο γίνεται πιο σύντομα και σήμερα θα ήθελα να σας καλέσω να έχουμε θετικό αποτέλεσμα για τον κανονισμό EBS και θα είναι αυτό ένα απαραίτητο βήμα για την ικανότητες της Ένωσης να κάνει, αυτό ακριβώς που μας, ρωτήσατε, που μας ζητήσατε. Ε, και θα κλείσει τώρα η συγγήτρια κυρία Μπελιέ. Δύο λεπτά παρακαλώ για να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν θα χρειαστώ δύο λεπτά. Νομίζω ότι η συζήτηση ήταν πολύ χρήσιμη και πλούσια. Ευχαριστώ τους κοιόδης συγητές. Θα ήθελα απλώς να τονίσω κάτι. Εάν η έκθεση έτσι όπως ψηφίστηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος αύριο και ενωθεί από το περιεχόμενό της, νομίζω ότι το θέμα της εντολής και το να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε μια διαπραγμάτευση ισορροπημένη, επικοδομητική με το Συμβούλιο θα πρέπει να την ξεχάσουμε ίσως, διότι ο στόχος είναι να επικυρώσουμε το πρωτόκολλο της ε, Ναγκόγια το σύντομότερο δυνατόν, διότι έχουμε, έχουμε όμως ευθύνη εξ ονόματος ε, των Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών συμφερόντων και όχι των εθνικών συμφερόντων ή κάποιου κλάδου φαρμακευτικού ή αγροτικού έχουμε το καθήκον και την ευθύνη να προωθήσουμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων και στην κοινή θέση που θα βρούμε με το Συμβούλιο και την Κομισιόν πρέπει να βρούμε μια θέση που θα είναι στο ύψος των προσδοκιών των Ευρωπαίων πολιτών, ούτως ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ωφέλη για ε, τους πολίτες και τους διάφορους ευρωπαϊκούς τομείς, διότι αδειάσουμε από το περιεχόμενό της την έκθεση δεν θα έχουμε αξιοπιστία και δεν θα μπορέσουμε να παρουσιαστούμε ε, στην διεθνή διάσκεψη στο τέλος του 2014. Επισύρω την προσοχή σας πάνω στο γεγονός αυτό και στην ψηφοφορία που θα λάβει η χώρα αύριο, ε, εφόσον η θέση της Επιτροπής Περιβάλλοντος συζητήθηκε ενδελεχώς και αποτέλεσε αντικείμενο συμβιβασμού. Θα προσθέσω απλώς ένα πράγμα. Όταν μιλάμε για νέες χρήσεις, δεν μιλούμε για αναδρομικότητα, δεν πρόκειται για αναδρομικότητα στην ψηφοφορία που είχαμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Είναι πληροφόρησα. ήμουν επίσης στην Αγκόγια και ξέρω ότι η εντολή που είχαμε για το Συμβούλιο και την Κομισιό με την Ένωση, την Αφρικανική, με τις τρίτες χώρες είναι να μην δεχτούμε την αναδρομικότητα. Δεν είμαι τόσο ασυνείδητη ώστε να εισαγάγω το θέμα αυτό και να έχουμε ε, μια νέα συζήτηση που θα μας κάνει να χάσουμε χρόνο. Δεν πρόκειται για αναδρομικότητα. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι τη στιγμή που θα εφαρμοστεί το κανονισμός και το πρωτόκολλο της Ναγκόγια θα υπάρχει ένας κανόνας για όλους τους Ευρωπαίους. Το θέμα των νέων χρήσεων είναι ένα θέμα ασφάλειας νομικής για να μπορέσουμε να ε, αποτρέψουμε στρεβλώσεις ανταγωνισμού μέσα στην Ένωση. Έχω ένα παράδειγμα και θα κλείσω με αυτό. Ας φανταστούμε ότι η Ένωση αποφασίσει να περάσουμε στα 110 χιλιόμετρα στους εθνικούς δρόμους και ε, αποφασίσουμε να περάσουμε μετά στα 60 διότι είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση και οι Ευρωπαίοι που θα έχουν αγοράσει ένα αυτοκίνητο ε, πριν τη ρύθμιση την ευρωπαϊκή θα μπορούν να τρέχουν με 110 χιλιόμετρα ενώ αυτοί που θα αγοράσουν νέο αυτοκίνητο μετά την ισχύ της ρύθμισης θα πρέπει να τηρούν τα 60 χιλιόμετρα. Έτσι είναι η περίπτωση αυτή. Ελπίζω ότι ήμουν αρκετά σαφής. Όταν μιλάμε για νέες χρήσεις, δεν πρόκειται για την εφαρμογή της πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για παλιές χρήσεις, ε, όταν θα ισχύσει ο κανονισμός θα πρέπει να ισχύει για το σύνολο ε, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με τρόπο δίκαιο και ισότιμο. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και αντίστοιχη ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα στρατηγική εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι της Επιτροπής Πολιτικών